Δεν έχουμε αρκετούς συναδέλφους για να ξεκινήσουμε, οπότε να περάσουμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε να ξεκινήσουμε απευθείας. Ανακοινώσεις της Προέδρους. Ενημέρωση για το διάλογο του ΠΑΚ. Δεν καταλήξαμε σε τελική συμφωνία για τη σχέδιο έκθεσης της κυρίας Φερέιρα αλλά η πλειοψηφία τη διαπραγματευτική ομάδα ζητά περισσότερα χέρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μορφή δήλωση από την πλευρά τη Επιτροπή για θέματα που έχει ζητήσει και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο 3 του σχεδίου έκθεση. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν οι διμερεί συζητήσει τι ερχόμενε ημέρε, προκειμένου να δούμε αν θα επιτελεστεί πρόοδο. Έχουμε μια ψηφοφορία πρώτα, το σημείο 5, ψηφοφορία για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ. Δεν είμαι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε κάρτες ψηφοφορίας. Ωραία. Καλύτερα να πάρετε τις κάρτες σας. I know uh, κύριος Λούντβιγκσον δεν έχει τη δική του.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 όλο δεν έχει την κάρτα του, ούτε ο Έντουαρτ. Έχουμε δύο παραπάνω στους σοσιαλιστές. Άλλος. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε τότε. Πρώτα απ' όλα συμβαστική α. Συμβαστική λύση α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική, ε και μπει σε δύο τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα προφορική τροπολογία των πρασίνων για την τροπολογία 32, όπου προστίθεται και το N, 42, όπου προστίθεται και το N private sector και ο ιδιωτικό τομέα. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 2α νέο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, C, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D, D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4α νέα προφορική τροπολογία των πρασίνων. Συμφωνούμε. Ωραία. Ψηφίσουμε με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56. Όχι, αυτή συμπεριλαμβάνεται στην προφορική. Συμβαστική ε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Όχι, όχι. Ξέχασα την F. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν θέλετε να ελέγξουμε. Πέρα της προφορίας. Ο που πήγε. Είναι ένας περισσότερος. Δίπλα στην κυρία Λούλη. 24 λοιπόν εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Με συγχωρείτε κατά τμήματα. Υπέρ, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές. Ας κάνουμε έναν έλεγχο για την 91. Ξαναπαντέ άπαντε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Νομίζω είναι 15 υπέρ, 19 κατά. Οπότε κερδίζουν οι 19. Ναι, αλλά και δύο ψήφου να είχαμε δεν θα αλλάξει το 19-15, οπότε και πάλι απορρίπτεται. 92 υπέρ. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. και πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 με προφορική τροπολογία των πρασίνων σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Συμφωνούμε με την προφορική τροπολογία. Ωραία. Πρώτο και δεύτερο τμήμα με την προφορική τροπολογία εννοείται. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 C την, με την 116 προφορική τροπολογία επίσης, συμφωνούμε. Υπάρχει καμιά αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ο έχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία στη δική του. Ψηφίζουμε λοιπόν την αρχική 116. 116 αρχική μορφή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας κάνουμε και έναν έλεγχο. Έχετε διαδικαστικό. Το μικρόφωνο σας. Ψηφίζουμε. Επειδή απορρίφθηκε η προφορική τροπολογία και επειδή χρειάζεται μία αντίρρηση για να απορριφθεί ούτως άλλως η προφορική, ψηφίζουμε την 116 χωρίς την προφορική τροπολογία. Του κυρίου Ραμόν Τεμόζα την, στην αρχική της μορφή, 116. Πέρας της πληροφορία. 25 προς 11. 13 δηλαδή με τις δύο επιπλέον ψήφους, οπότε εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 125 Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. 16 προς 20. Οπότε απορρίπτεται. Ακόμη και αν ήταν 18. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, ας κάνουμε έλεγχο. Σοσιαλιστές. Ωραία, πέρα της ψηφοφορίας. 20 προς 16, δηλαδή 20 προς 18 με τις δύο πλεονάζουσες ψήφους με τις δύο επιπλέον μάλλον ψήφους. Οπότε και πάλι εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Δεκαπέντε με προφορική τροπολογία. Συμφωνούμε με την προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Οπότε με την προφορική τροπολογία όπως τροποποιήθηκε η τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σύγχυση. Ας ψηφίσουμε. Εψήφισαν πάντες πέρας. Σύγχυση, σύγχυση στο ΕΛΚ. Κοιτάξτε, τι ψηφίζουμε, την προφορική τροπολογία ή το αρχικό κείμενο. Ψηφίζουμε το κείμενο όπω τροποποιήθηκε, διότι δεν υπήρξε αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Θέλετε να ψηφίσουμε και την προφορική τροπολογία. Ωραία. Προφορική προφολογία αλλάζω τον όρο austerity με consolidation. Συμφωνούμε. Θέλουμε, θέλετε να ξαναψηφίσουμε. Ωραία. Άκυρη η πρώτη ψηφοφορία. Ξαναψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 15 με την αλλαγή του austerity σε consolidation. Υπέρ. Ας αρχίσουμε. Πέρας. Εντάξει. Πέρας. Νομίζω ότι εγκρίθηκε αυτή τη φορά. 27 προς 1. Οπότε μια χαρά. Κυρία Πρόεδρε, είμαι πολύ υπάκος. Διαβάζω τι λέει το έγγραφο και βλέπω ένα μείον. Αυτό κατάλαβα. Νομίζω τα καταφέραμε τελικά. Δεν καταγράφηκε. Τη λογική σκέψη C, 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο. Δεν χρειάζεται 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω, Πολ, πάλι έχασες τη σειρά. Η υπόλοιπη ομάδα σου ε, ψήφισε το αντίθετο. Κοιτάξτε, κάνουν ε, ακριβώς ό,τι και στο ΙΟΜΠ στο κόμμα της Γαλλίας. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, όχι. Απεπτή. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το κείμενο πώς τοποποιήθηκε ηλεκτρονικά. ψήφους εγκρίνεται 32 υπέρ, 1, μία ψήφος κατά, άρα 34 υπέρ, μία ψήφο κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Um, Would, those who are leaving do so quickly and... Παρακαλώ γρήγορα να αποχωρήσετε και αθόρυβα για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε με την έκθεση του Έντουαρντ. No, it's okay. Okay, um, Ας ε, προχωρήσουμε. Ησυχία παρακαλώ για να μπορέσει και ο Έντουαρ να μιλήσει. Ευρωπαϊκές στατιστικές. Εξέταση των τροπολογιών για την έκθεση του Έντουαρτ Σικλούνα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε για ποιο λόγο καλούμεθα να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Το βασικό γεγονό που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και γεννά ερωτηματικά σε σχέση με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων ναι, ήταν, όπω όλοι γνωρίζουμε, τα περιστατικά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Έχουμε δε και τα πακέτα των 6 και των 2 νομοθετημάτων, six packs και two pack, που βασίζονται σε στατιστικούς δείκτες για καθοδήγηση, για λήψη αποφάσεων, για επιβολή κυρώσεων και το καθεξής. Πολύ μεγάλο άχθος λοιπόν, πολύ μεγάλη πίεση για τους δείκτες Διότι πρέπει να ξέρουμε τι πραγματικά ισχύει, όχι τι φαίνεται να ισχύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εξετάσαμε την πρόταση, κρίναμε ότι ήταν ιδιαίτερα δύναμη, ακόμη και ε, στα εκτιμώντα, στις αιτιολογικές σκέψεις. Πρέπει να καταδείξουμε πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο είναι όντως σημαντική αυτή η έκθεση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα παρελθόντα περιστατικά που ήταν και μια ε, που ήταν ε, μία από τις αιτίες ε, μιας τεράστιας κρίσης και καλυμμένης για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της παραποίησης των στατιστικών στοιχείων. Εξέτασα τις διάφορες τροπολογίες και σαφέστατα τροφοδοτούν τη συζήτηση και τις διαπραγματεύσεις Μπορώ να δεχτώ τις περισσότερες από αυτές. και δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα να καταλήξουμε σε μια συμβαστική διατύπωση για τι διάφορε αυτέ τις τροπολογίες. Κάτι άλλο που τόνισαν ιδιαίτερω και οι σκιώδει καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία είναι ο δημοκρατικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκό καθώ και σε εθνικό επίπεδο για να νομιμοποιήσει τη διαδικασία και να διατηρήσει τον έλεγχο. Καλωσορίζω και αυτή την παρατήρηση των σκιωδών. Μία πτυχή που φαίνεται τεχνική πλην όμως έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η εξή. Ε. Θα πρέπει να διατηρηθεί μια καλή ιδιαιτερη σημασια ειναι η εξης θα πρεπει ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκά συστήματα, το ESB, e στατιστικό σύστημα της ΕΚΤ και το δίκτυο των ε, εθνικών στατιστικών υπηρεσιών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ESS, ούτως ώστε να, μην, να αποφύγουμε την επικάλυψη κατά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και να αλληλοσυμπληρούνται οι δύο οργανισμοί. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση του ελέγχου των στατιστικών στοιχείων και της εμπιστευτικότητας των στατιστικών ε, στοιχείων τους. Ε, το θέμα του αν είναι και φιλικά προς το χρήστη τα στατιστικά στοιχεία πάντοτε ανακύπτει. Ε, εάν συλλέγονται τα στατιστικά στοιχεία αλλά δεν διαδίδονται, κοινοποιούνται με ένα φιλικό προς το χρήστη τρόπο, τότε δυσχεραίνεται η πρόσβαση. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν περιπλοκές και να εξασφαλίζεται μια εύκολη πρόσβαση σε μια εποχή όπου πολλοί έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, τονίστηκε ε, ε, η σημασία της ανεξαρτησίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, του Eurostat δηλαδή, καθώς και των Εθνικών Στατιστικών Ιδρυμάτων. στο παρόδο, ναι μεν, χρειαζόμαστε την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των ε, στατιστικών οργανισμών, όμως ε, αυτό συνεπάγεται τροποποίηση της νομοθεσίας που να προβλέπει ρητά αυτή την ανεξαρτησία και να είναι και ουσιαστική. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Κάποιες χώρες έχουν ε, ήδη επιτύχει να υιοθετήσουν υψηλότατα πρότυπα ανεξαρτησίας για τα εθνικά στατιστικά σου ιδρύματα, άλλες πάλι όχι. Ε, σε κάποιες χώρες ε, υπάγονται ε, σε ένα υπουργείο και άρα λογοδοτούν στον εκάστοτε υπουργό. Ε, δημιουργούνται μεγάλες συγκρούσεις συμφερόντων με τα αναμενόμενα κακά αποτελέσματα. Προσπαθήσαμε στις τροπολογίες που θα εξετάσουμε, στο προηγούμενο σχέδιο δηλαδή, να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα αφενό στη Eurostat και αφετέρου τα εθνικά στατιστικά ιδρύματα σε σχέση με τι απαιτήσει μα ε, προ αυτά. Ε, Ποιε πρέπει να είναι αυτέ. Στο ιδανικό σενάριο θα έπρεπε να λογοδοτούν όχι ε, στην κυβέρνηση ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίως τα εθνικά στατιστικά ιδρύματα θα έπρεπε όταν διορίζεται ο επικεφαλής Φερρυπίν να εξετάζεται την υποψηφιότητά του από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το ίδιο ε, και για τη γύρω Το επικεφαλής της αρμόδιας ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, θα έπρεπε να εξετάζεται και να χορηγείται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε όμως να ζητήσουμε τροποποίηση της συνθήκης. Ε. Θα πρέπει να αναμείνουμε μια τροποποίηση συνθήκης, μάλλον αν πραγματικά θέλουμε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα να συνάδει με το Στατιστικό Πρόγραμμα της ΕΚΤ. Μπορεί κάποιοι να μας πούν για ποιο λόγο το ζητάτε αυτό, να μπορούμε να ζητήσουμε από οποιονδήποτε επίτροπο να, αυτήν την ίδια ανεξαρτησία. Ζητήσαμε και κάποιες χώρες ζητούν όντως να υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία προς το στατιστικό πρόγραμμα της ΕΚΤΕ. Οι δείκτες όμως που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως ε, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την επιβολή κυρώσεων, πρέπει να είναι αντικειμενικά αληθή τα στοιχεία, να εκλείψει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και γι' αυτό ζητούμε αυτή την ανεξαρτησία, όπως και για τις, Ευρωπαϊκές Κεντρικές, ε, τις Εθνικές ε, Κεντρικές Τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, αλλά ακολουθούμε αυτό τον προσανατολισμό. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε κάποιες τροπολογίες που σχετίζονται με τις επικυρώσεις και τα πρόστιμα για την ε, παραποίηση και το μαγείρεμα των στατιστικών στοιχείων. Ας μην μιλάμε για την ιστορία, ας μιλήσουμε για το μέλλον. Και ε, ο μόνος τρόπος είναι να εισαγάγουμε κυρώσεις και πρόστιμα, ούτως ώστε ποτέ κανείς στο μέλλον να μην έχει τη δυνατότητα να παραποιήσει εκ νέου στατιστικά στοιχεία. Η Σάρον κατέθεσε μια κατεμή ενδιαφέρουσα τροπολογία ένα μοντέλο που εμφαρμόζεται ήδη στη Eurostat, δηλαδή να εφαρμοστεί και στο εθνικό επίπεδο ε, με ένα εθνικό συμβουλευτικό όργανο για το Εθνικό Στατιστικό Ίδρυμα. Αυτό υπάρχει σε κάποιες χώρες, στη δικιά μου παραδείγματος χάρη υπάρχει, αλλά όχι σε όλες. Αναμένω τώρα τα σχόλια των σχεδόν. και προσβλέπω στην ε, σύσκεψη που θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στο τελικό συμβαστικό κείμενο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκπροσωπεί κάποιος τον Ζαν Πολ ή το ΕΛΚΑ γενικότερα. Όχι, τότε η Σοφή είναι η επόμενη σκιώδηση συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Οφείλω να πω ότι διάβασα όλες τις τροπολογίες και την έκθεση και έχω ανησυχήσει λίγο, έχω θορυβηθεί. Γιατί ε, μιλούμε για την ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών ή αρχών και της Eurostat και τελικά πού θα καταλήξουμε. Ε, η Eurostat είναι ένα συνοθήλευμα ε, κανόνων ε, εκεί που ισχύει για ε, τη λογοδοσία και την ευθύνη. Και πώς κανονίζεται την ανεξαρτησία της Eurostat, όχι μόνο τις διαδικασίες του διορισμού, αλλά και είπαμε ότι ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και τελικά ουσιαστικά είναι υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι και αλλιώ. Και ισχύει ο κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Εσείς ο ίδιος προτείνετε να περιοριστεί το περιθώριο χειρισμών ε, που έχει ε, το όλο στατιστικό σύστημα ότι διαχωρίζεται ε, από το σύστημα κεντρικών τραπεζών. Υπάρχουν τροπολογίες που ζητούν να δημιουργηθεί ένα είδος εποπτικού συμβουλίου που μπορεί ως ιδέα να είναι καλό, αλλά μετά αυτό Πώς θα συνάδει με τον εποπτικό ή ελεκτικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων ή το δικό μας. Υπάρχουν τροπολογίες που ζητούν ένα είδος πιστοποίησης ε, και ε, των ε, στοιχείων από το ελεκτικό συνέδριο. Είναι λοιπόν αυτό ένα μπέρδεμα και στο τέλος δεν καταλαβαίνω ποιος θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος και πώς θα το λύσουμε αυτό χωρίς να ζητήσουμε αναθεώρηση των συνθήκων. Και βέβαια χρειάζεται να βρούμε λύσεις, αν ε, δεν αναθεωρηθεί η συνθήκη, αλλά ανησυχώ πραγματικά για το που θα βγάλει αυτή η ιστορία. Και για τα πρόστιμα που συνδέεται και αυτό, ξέρω ότι είναι τρεις οι εναλλακτικέ λύσεις. Εσείς προτείνετε τα πρόστιμα να αποφασίζονται από το Συμβούλιο. Ειλικρινά την τελευταία δεκαετία είδαμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Αν τα κράτη-μέλη ε, ελέγχουν το ένα το άλλο, ουσιαστικά δεν το κάνουν ποτέ. Κανονικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει για τα πρόστιμα. Η πράσινη, ο Φιλίπ Λαμπέρτς πρότεινε ένα ενδιάμεσο σύστημα να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποφασίζει το Συμβούλιο με ε, αντίστροφη ειδική πλειοψηφία. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ να εκφράσω την ανησυχία μου. Γιατί είναι περίπλοκο το σύστημα και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Thank you. Next it's Yes, thank you, Sharon. Ο Φίλιπ Λάμπερτ, Ευχαριστώ, Σάρον. Δεν ξέρω τώρα εγώ τι να πω. Πρέπει να συμπεράνω από την προσέλευση των συναδέλφων όταν συζητούμε τις στατιστικές ότι ενδιαφερόμαστε μόνο λίγοι σε πολιτικές που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Ελπίζω όχι. Απλώς το εκλαμβάνω ως εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και στην ποιότητα της δουλειάς μας. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε μερικά στοιχεία. Δεν θα επαναλαμβάνω κάθε φορά ότι συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση όσο και το ύφος της έκθεσης του εισηγητού. Δεν υπάρχουν πολλά τα σημεία διαφωνίας για την ανεξαρτησία των επικεφαλής των εθνικών στατιστικών ε, ε, υπηρεσιών. Νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο και ίσως εκεί να διαφωνήσω μαζί σου. Αυτό που μετράει κανείς είναι αυτό που παίρνει ως στοιχεία ή προσπαθεί να συλλέξει. Και το να αποφασίσει τι στατιστικά στοιχεία θα συλλέξει είναι πολιτική απόφαση. Δηλαδή, αν αποφασίσει μια κοινωνία ότι είναι σημαντικό να μειώσει ε, το οικολογικό της αποτύπωμα ή να μειώσει ε, τις ανισότητες στο εισόδημα, μπορεί να αποφασίσουν ότι χρειάζεται να το μετρήσουν. Δεν θα το αποφασίσει αυτό ε, η στατιστική υπηρεσία. Μπορεί να έχει ε, ανεξαρτησία στις μεθόδους που θα ακολουθήσει τις επιστημονικές και σε ποιο βαθμό ε, και με ποιο τρόπο θα στηλέξει τα στοιχεία, αλλά δεν είναι πολιτικό σώμα για να αποφασίσει ποια στοιχεία θα συλλέξουν. Εγώ είμαι ακρεφνής υποστηρικτής της ε, ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και θα το κάνω και για τη στατιστική υπηρεσία, αλλά τις πολιτικές αποφάσεις δεν τις παίρνουν ε, ε, στατιστικές αρχές, αλλά ερετοί, άνθρωποι δηλαδή. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τη χρυσή τομή ανάμεσα στη λογοδοσία και στην ανεξαρτησία αλλά και τη δημοκρατική νομιμότητα. Δηλαδή, αυτοί που εργάζονται και στι κεντρικέ τράπεζε και στατιστικέ υπηρεσίε δεν είναι τέλειοι, ούτε άγιοι είναι οι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι και με πολιτικέ απόψει και με προκαταλήψεις όπω όλοι μα. Δεν είναι καλύτερη ποιότητα, καλύτερη πάστας άνθρωποι. Για το Γενικό Διευθυντή θα ήθελα μόνο να πω ότι... Ε, για το θέμα του φίλου εκφράσαμε κάποια ευαισθησία και θέλω να το χρησιμάσετε. Για την αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ευχαριστώ Σοφή που με υποστηρίζεις για τις κυρώσεις κατά πρόστιμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας λογικός συμβιβασμός. Αυτά. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Okay, Η Βίκη δεν είναι εδώ από το ECR, ούτε, ούτε η γκουε εκπροσωπείται, εγώ μένω μόνο. Γιατί κατέθεσα και εγώ κάποιες τροπολογίες. Αυτές οι τροπολογίες προέκυψαν από τη συζήτηση που έκαναμε με τον Τόμας Βάισε, τον πρόεδρο της ΕΣΚΑ, όταν ήρθε στην ακρόαση. Ε, δυστυχώς ε, δεν ήταν άθροα η προσέλευση. Το καλό είναι ότι ακριβώς ε, Γι' αυτό το λόγο μου μας έδωσαν διεξοδικές ε, διευκρινήσεις ε, για διάφορα σημεία και πρότεινε κάτι πολύ σωστό και έκρινα εγώ ότι υπό τη μορφή τροπολογίας έπρεπε να το συμπεριλάβουμε μέσα στο κείμενο ε, και σχετίζονται αυτό με την, τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, ξυπακούεται όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά κάποτε στις χώρες κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης υπήρχε μια τάση οι γυναίκες να είναι επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Ιδρυμάτων. Μετά την προσχώρηση των χωρών εξέλιψαν οι γυναίκες αυτές. Ε, πολύ περίεργο, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό το λόγο θεώρησα ότι άξιζε να το τονίσουμε αυτό το στοιχείο. Ξέρετε ότι τα μαθηματικά και τα στατιστικά, η στατιστική δεν μπορεί να είναι ένας τομέας όπου υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες λόγω μόνο της έλλειψης ακαδημαϊκών πτυχίων κτλ. Λοιπόν, είναι αυτονόητε οι τροπολογίε, όπω έλεγα. Το περιεχόμενό του είναι αυτονόητο και μάλλον θα το δεχτεί ο εισηγητή, το ελπίζω. Ο στόχο είναι να είναι ασφαλέστερα τα στατιστικά στοιχεία και να μην μπορούν να χειραγωγούνται από ε, τους πολιτικούς. Δεν θα πω τίποτα άλλο για να ε, προωθήσω τις τροπολογίες μου. Ε, εκπροσωπείται και η Eurostat εδώ, βλέπω, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω το ηχηρό πολιτικό μήνυμα που η έκθεση αυτή αποστελεί, η έκθεση του κυρίου Σουκλούνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να ενισχύσουν το σύστημα και την διακυβέρνησή του. Από αυτήν την άποψη η προστασία και η ενίσχυση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας είναι καθοριστική σημασία στην γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του ευρωπαϊκού και εθνικού επίπεδου. Η δημοκρατική λογοδοσία είναι επίσης ένα θέμα που μας απασχολεί. Είναι ζωτική σημασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χαρά θα στηρίξει όλες τις τροπολογίες που συμπεριλαμβάνει η έκθεση. Επίσης, ο συστηματικός στατιστικός διάλογος είναι κάτι που υποστηρίζουμε συμπληρώνοντας κάτι που ήδη γίνεται σε έναν βαθμό στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών. Ήδη κάποια από τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικά. Η ακρόαση του Γενικού Διευθυντή στην Επιτροπή σας ήταν ήδη ένα δείγμα και το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Επίσης, συμφωνούμε ότι η πολιτική ίσων ευκαιριών θα πρέπει να εφαρμοστεί ενώ σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, της κυρώσεις. Αυτό είναι ένα σχετικός νέο στοιχείο στον τομέα της στατιστικής, αλλά και πάλι είμαστε υπέρ της αρχής αυτής. Κατά την άποψή μας όμως, θα πρέπει να στοχεύσουν αυτές οι κυρίως αυτά τα πρόστιμα τους τομείς της στατιστικής που είναι άκρας σημασίας. Στατιστικά στοιχεία λόγου χάρη για τα δημοσιονομικά για τις διαδικασίες EDP, για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, για το υπερβολικό έλλειμμα. δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια γενική αρχή που να διέπει όλο τον τομέα της στατιστικής. Θα πρέπει να, να εντοπίσουμε τα σημεία που αυτό θα είναι εύστοχο, που θα έχει νόημα και θα είναι και εφικτό. Διότι σημαίνει ότι θα χρειαστούν και επενδύσεις από την πλευρά της Eurostat και δεν έχουμε επαρκείς πόρους για να αναλάβουμε τόσο μεγάλο έργο για όλων των ειδών τα στατιστικά στοιχεία. Νομίζω η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εύρωστη διαχείριση ποιότητας πολιτικής ποιότητας είναι η κατεύθυνση που και εμεί θέλουμε να ακολουθήσουμε σε τομείς που ακριβώς χρειάζεται τέτοια διαχείριση αλλά όχι αδιακρίτως σε όλους τους τομείς της στατιστικής. Εκεί που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες χρήσεις. Το τρίτο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, αφορά την τροπολογία της Προέδρου που αφορά την ε, δημιουργία φορέων στατιστική σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι που νομίζουμε ότι θα συμβάλλει στην εναρμόνιση των διατάξεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ μπορεί να υπάρχει και μια ευκαιρία να εγκαθιδρυθεί ένας συσχετισμός, γιατί χρήσιμο θα είναι αυτή η εθνική φορείς των εθνικών στατιστικών ε, υπηρεσιών να καλύψουν τα κενά. Θα μπορούσε να υπάρχει λοιπόν μια παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του θέματος αυτού και να ευθυγραμμίσουμε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Έντουαρτ. Ευχαριστώ επειδή γενικώ υπήρξε συμφωνία για πολλέ τροπολογίε, να σταθώ σε όσα σημεία υπήρξαν διαφωνίε, ιδίω με τον κύριο Λάμπερτ, όπου συζητήσαμε το πόσο οι εθνικέ υπηρεσίε θα πρέπει να είναι ανεξάρτητε. Νομίζω είναι θέμα ερμηνεία τη ανεξαρτησία. Δεν μιλάμε για πολιτική ανεξαρτησία. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία στο Κοινοβούλιο. Και για το σχόλιο που ακούσαμε τώρα από την Επιτροπή για την τροπολογία τη κυρία Μπόλ, θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος συμβουλίου, συμβουλίου αυτών των ε, φορέων, όπου να υπάρχει λογοδοσία για το έργο των ε, υπηρεσιών, των στατιστικών υπηρεσιών. Έτσι, κακώ φοβάται ο κύριο Λάμπερτ ότι κάποια δεδομένα μπορεί να μην ε, συλλέγονται. Όχι, θα καλύπτονται όλα. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών, εγώ θα προτιμούσα έμφαση να δοθεί στο εθνικό επίπεδο. Διότι εκεί είναι η πηγή των προβλημάτων, εφόσον εκεί συλλέγονται τα δεδομένα σε πρώτη φάση. Είμαστε αυτό που τρώμε, λέμε. Το ίδιο και για, τα, για, τα, για τις υπηρεσίες. Δηλαδή, όπως και στους υπολογιστές. Υπάρχει ο κάδος απορριμμάτων. Εδώ λοιπόν Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ένα σχετικό συντονισμό. Όμω ε, οι υπηρεσίε δεν θα πρέπει να είναι υπόλογε σε έναν ε, υπουργό που να αποφασίζει πότε θα δημοσιεύονται τα στατιστικά στοιχεία σε προεκλογική περίοδο ή αν θα υπάρξει τρίμερη καθυστέρηση ούτω καθεξή. Αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί στο παρελθόν και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν. Θέλουμε να ενισχυθούν οι εθνικέ στατιστικέ υπηρεσίε. Να είναι ανεξάρτητε ω προ το διορισμό των επικεφαλή των διευθυντών, τα κονδύλια με τα οποία θα πρικοδοτούνται αλλά να λογοδοτούν στα εθνικά κοινοβούλια. Όπω θα θέλαμε να συμβαίνει και με τη Eurostat. Η Σόφη ανέφερε κάτι που και εμένα με προβληματίζει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τόσο όσο θα θέλαμε και να φτάσουμε και σε αλλαγή τη συνθήκη. Χωρί να φτάσουμε και σε αλλαγή τη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε και τις προτάσεις. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να επιτελέσουμε πρόοδο εδώ. Και αν συναντηθούμε στο Στρασβούργο με τους σκέδους συζητητές, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Η ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για τη 17 η Δεκεμβρίου και ελπίζουμε το Μάρτιο να ψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Δηλαδή ελπίζουμε να συμφωνηθεί μέχρι τότε. Να έχουμε καταλήξει. Ευχαριστώ όλους. Και προχωρούμε στο σημείο 4 της ημέρας της Η κυρία Νετφέλτ το λόγο, δεν την έχει δει η πρόεδρος. Σόφη. Ε, πριν πάμε στο Στρασβούργο σε ψηφοφορία, δεν θα ήταν ε, σκόπιμο να έχουμε μια γενική επισκόπηση, ένα πίνακα ενδεχομένω. Γιατί είναι τόσο πολλές διαφορετικές οι προτάσεις ε, για την εποπτεία, για τη λογοδοσία, για το ποιος αποφασίζει τι. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια συνολική εικόνα των διαφόρων ε, δυνατοτήτων ρυθμίσεων για να μην υπάρχει επικάλυψη ή ακόμα και σύγκρουση στις ρυθμίσεις που αποφασίζουμε. Και για τη λογοδοσία του επικεφαλής της Eurostat και των Προέδρων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Μα, Σόφη, δεν ψηφίζουμε την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο, την Δευτέρα στις 17. Όταν όλοι θα θέλουν να έχουν ήδη φύγει για διακοπές, ελπίζουμε να μην έχουν φύγει. Στις 17, όχι την άλλη εβδομάδα. 17 και 18 Δεκεμβρίου. Το σημειώνουμε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Um, okay, moving on now to point which is an agenda for Πάμε στο σημείο 4. Ατζέντα για επαρκή λέει ασφαλή και βιώσιμε συντάξει. Είναι η έκθεση του κυρίου Τόμας Μαν. Θα του δώσω το λόγο. Äh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητή Σάρων. Έχω κάνει μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης. Είναι η έκθεση πρωτοβουλίας εκεί, όπου συμμετέχω κι εγώ, είμαι μέλος και καλό είναι να γνωμοδοτήσει και η Οικονομική Επιτροπή, γιατί έχει τις δικές της προτεραιότητες. Έχουμε εδώ τρεις πυλώνες ε, του συνταξιδοτικού, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι βασικές συντάξεις, οι κύριες λεγόμενες. Έχουμε εμπειρία στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εκεί να τηρηθεί ε, απ' έξω ταπεινά για την αρμοδιότητα των κρατών μελών, να κάνετε κριτικές αναλύσεις. Και σε χώρες που δεν έχουμε ε, διανόμου επιβολή βασικής σύνταξης, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε για να καλύψετε τα κενά. Ε, τα συστήματά μας θα πρέπει να αντέχουν στη δημοκρατία και στη δημογραφία. Ε, για το δεύτερο να χαίρομαι πολύ γιατί έχουμε τώρα ίδιες εξουσίε και αρμοδιότητε και να ευχαριστήσω τη Σάρεν Μπόλ ιδιαίτερα για ε, τη συνεργασία και την υποστήριξη. Ε, η έκθεση είναι έξι σελιδούλε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε αγαπητοί συνάδελφοι ότι διάβασα καμιά εικοσαριά συστήματα ε, των κρατών μελών, 300 με 400 σελίδες που χρειάστηκε να συνοψίσω. Είναι πολύ διαφορετική εμπειρία στα κράτη-μέλη και σε πολλές χώρες. Ε, έχουμε βέβαια υποστήριξη για τα εκάστοτε συστήματα, αλλά ορισμένα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα σωστά συστήματα, είναι τα κατάλληλα, αντέχουν στο μέλλον. Λοιπόν, σε αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχουμε από τι διάφορε πρωτοβουλίε, οι τομεί που μα αφορούν εμά είναι η πρωτοβουλία επαριθμών 9 για τι κατάλληλε ε, συντάξει και η οδηγία ε, IORP, η φερικιότητα 2, η πρωτοβουλία 12 και η 13 τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συντάξεων Παροχών. Το 18 αφορά τους φόρους και το 19 την ασφάλεια ζωής και χαίρομαι που έχουμε αρμοδιότητες και θα πρέπει όλοι να συντονιστούμε οπωσδήποτε. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να φροντίσουμε, να προσέξουμε οι διαφορετικότητες των κρατών μελών να λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σύστημα να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πρωτοβουλία υπαριθμών 11. Απορρίπτει τη ρυθμιστική εναρμόνιση των ποσοτικών ή ποιοτικών διασφαλίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διαχείριση κινδύνου ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ε, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ελευθερία και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ε, οι συνάδελφοι σε μεγάλο βαθμό. Ο πυρήνας όμως της έκθεσης είναι η απόρριψη των ποσοστώσεων ιδίων κεφαλαίων και η αναθεώρηση της οδηγίας για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συντάξεων Παροχών. Και έρχομαι τώρα στη φεραγιότητα 2, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Και βέβαια θέλουμε οι εταιρείε να ε, είναι εξασφαλισμένες και με ίδιο κεφάλαιο για το μέλλον. Αλλά όταν μας λένε ότι θα πρέπει να ε, μεταφέρουμε εδώ την εμπειρία που έχουμε από τις ασφάλειες ζωής και από άλλους τομείς. Μα αυτά τα πράγματα δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Τι εμπειρίες έχουμε. Είναι κάπως διαφορετικές αυτές. Παράδειγμα, ειδικέ συντάξεις των επιχειρήσεων. Αυτά είναι κοινωνικά συστήματα εθελοντικής βάσης σε πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχουν δυνατότητες να έχουν λόγο και οι κοινωνικοί εταίροι. Στην ασφάλεια ζωής αυτό δεν ισχύει. Ας πούμε, έχουμε στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, ε, ένα ε, πολύ καλό σύστημα ε, συνταξιδοτικό επικορικό και έχουμε περάσει τη μεγαλύτερη κρίση, ναι, την έχουμε περάσει και έχει αποδειχθεί η σταθερότητα αυτών των συστημάτων και αυτή την εμπειρία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Ποια, ποιο είναι η κίνδυνη όταν έχουμε συστήματα που λειτουργούν σωστά και προτείνονται νέες ποσοστώσεις ιδίων κεφαλαίων, υπάρχει ο κίνδυνος, επαναλαμβάνω, συστήματα που λειτουργούν σωστά, ξαφνικά να με τέτοιο κόστος που θα έχουν επιπτώσεις. Δηλαδή είτε θα μειωθεί η σύνταξη ε, ε, των εργαζομένων, είτε θα καταργηθούν αυτά τα συστήματα που έχουν οι εταιρείε για την ασφάλιση των εργαζομένων τους, πέρα από τη βασική σύνταξη. Αυτά είναι σωστά ε, συστήματα υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των εργοδοτών και δεν μπορεί η Ευρώπη να τα καταργήσει έτσι. Είναι λάθος μήνυμα ή να τα διακυβεύσει. Τον Απρίλιο του 2011 και τον Ιούνιο του 2012 και η ΕΤΟΚ, δηλαδή τα συνδικάτα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, αλλά και η Business Europe που είναι οι εργοδότες, από κοινού ε, συνέταξαν μία επιστολή και είπαν για τη φερεγγιότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί σε συντάξει γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και είναι το πιο λάθος μήνυμα που μπορεί κανείς να στείλει. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία παριθμών 11. Άλλο θέμα, η πρωτοβουλία παριθμών 17. Ε, καλωσορίζω και χαιρετώ την πρόταση να έχουμε ε, ε, σχέδια σύσταση διασυνοριακών υπηρεσιών καταγραφής για το δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να είναι και φθηνό, χωρίς επαχθείς νομικές και διοικητικές δικασίες. Στην τρίτη στήλη, στις ιδιωτικές συντάξεις ή στις συντάξεις των εταιριών, δεν θα πρέπει να καταργηθεί ε, ο πρώτος πυλώνα στις βάρους του τρίτου πυλώνα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα με ειφορία, με ε, βιωσιμότητα και για τον τρίτο πυλώνα και αξιοπιστία. Και ποια είναι η νομική βάση, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί στη Λευκή Βίβλο δεν βλέπω και πολλά πράγματα σχετικά. Διαπιστώνω ότι τα συστήματα μας κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίση. Στην πρωτοβουλία υπάρχουν 13 υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εθελοντικούς κωδικές στον πληθυντικό συμπεριφοράς για τον τρίτο πυλώνα. Αυτή η μανία επιτέλους για ρύθμιση κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ε, εντάξει, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, συμφωνώ, να κοιτάξουν ε, να ανταποκριθούν στο καθήκον που έχουν, να εξασφαλίζουν σύνταξη για τους πολίτες. Αλλά όχι με αυτή τη μανία για υπερρύθμιση όλων. Να απευθύνουμε πήγους έγκληση στα κράτη-μέλη να αναλάβουν ρυθμιστική δράση. Ωραία. Αλλά μέχρι εκεί. Ελπίζω να σας κάλυψα και θα παρακαλούσα σε συνεννόηση με τους κοιόδες ηγητές να έχουμε μια ισόρροπη έκθεση και να μπορούμε να πούμε και στους εργοδότες και στους εργαζομένους ότι θέλουμε ένα σύστημα ε, επιχειρησιακών συντάξεων που να μπορεί να χρηματοδοτείται και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζω από κοινού να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμφιβασμό. Ευχαριστώ και πάλι την Πρόεδρο. Και ε, σας ευχαριστώ που μας επιτρέψετε να πούμε ότι έχουμε ίδιες αρμοδιότητε εδώ στην Οικονομική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλε τώρα από πλευρά των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχίζοντας να ευχαριστήσω τον Τόμας Μάνε. Πραγματικά ήταν διεξοδική και ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της έκθεσης. Ε, είναι καταπληκτικό επαλτήριο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις μας. Είμαι πεπισμένος ότι θα είναι επικοδομητική όλη η διαπραγματευτική διαδικασία για το γενικό ζήτημα των συντάξεων τώρα. Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για να βρούμε σωστές αποχρώσεις για τα επιμέρου ζητήματα ε, επί της ουσίας πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα όταν μιλάμε για συνταξιοδοτικά συστήματα και αυτό θα πρέπει να το σεβαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της συνταξιοδότησης. Παραδείγματος χάρη, προσαρμογή των συντάξεων, ε, μεταφορά των συντάξιμων δικαιωμάτων για να κατοχυρωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, επίση να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου ή ηλικία, ε, ενίσχυση τη προστασία των καταναλωτών ε, και βελτίωση του κλίματο εργασία. Υπάρχουν και διάφορα άλλα συναφή σημεία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η γενικότερη τάση θα έπρεπε να είναι ένας συνδυασμός του πλήρου σεβασμού της εθνικής αρμοδιότητας ε, και μια ρεαλιστικής προσέγγισης και συνεργασίας στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων, γιατί σαφέστατα μπορεί να προσφέρει την αξία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τώρα ασχοληθούμε με επιμέρους ζητήματα της πρωτοβουλίας της Λευκής Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να κάνω κάποια προκατακτικά σχόλια. Πρώτον, σε σχέση με τις επαγγελματικέ ε, συντάξεις. Ε, μιλάμε για την αύξηση της ηλικία ε, συνταξιοδότησης. Είναι αναφυσβήτητο ότι πρέπει να θεσπίσουμε μια υψηλότερη συνταξιδοτική ηλικία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι βιώσιμο το νέο σύστημα σε σχέση με την προηγούμενη ηλικία συνταξιοδότησης. θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμο ένα συνταξιοδοτικό σύστημα ε, όταν αποχωρούμε υπερβολικά νωρί από την ενεργό ζωή. Θα πρέπει επίση να συνυπολογιστούν διάφοροι παράγοντε, όπω παραδείγματο χάρη το αυξημένο προσδόκιμο ζωή και τα νέα δημογραφικά δεδομένα. Αποκλείται να επιτύχουμε ένα επαρκέ, βιώσιμο και ασφαλέ συνταξιοδοτικό σύστημα, εάν δεν επικρατήσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην αγορά εργασία και καλύτερη αποτίμηση ε, της ε, ενεργού ζωής και της ε, υπόλοιπης ζωής μετά τη σύνταξη. Ε, η Ευρωπαϊκή Οδηγία σε σχέση με τα επαγγελματικά συνταξιδοτικά συστήματα έχει μεγάλη σημασία για τα ποσοτικά ζητήματα, δηλαδή για τις ε, επαγγελματικές συντάξεις. Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού και δημιουργούνται προβλήματα διότι ε, το κάθε ένα συνεπάγεται διαφορετικό κόστος και άρα πρέπει να προσέξουμε ως προς την νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτό το στάδιο θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε ασφαλείς συντάξεις ε, και άρα ε, η ανάλυση, η ποσοτική ανάλυση των διαφόρων εναλλακτικών συστημάτων έχει καταλητική σημασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντατικοποιεί τις εργασίες της σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα, με τις ατομικές δηλαδή συντάξεις. Όντως θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων που έχουμε καθώς και να ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να ε, προστατεύσει και το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τι υποχρεωτικέ ε, συλλογικέ συντάξει, γιατί όταν ο εργοδότη είναι αφαιρέγγυο πλέον δεν κατοχυρώνεται ο δεύτερο ε, πυλώνα. Εν τέλει, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβάλλει και να προωθήσει την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα, καθώ και τη παρακολούθηση των επαγγελματικών συντάξεων. Είναι κατεπήγον λοιπόν να συντονίσουμε όλα τα εθνικά συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτύχουμε αποτελεσματικό έλεγχο των επαγγελματικών συντάξεων. Αφήστε που κατά τη διάρκεια τη επαγγελματική του ζωής ε, πολλοί εργάζονται σε διάφορα κράτη-μέλη της Ένωση. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των συντάξιμων, κατοχυρωμένων συντάξιμων δικαιωμάτων του. Ε, μόνο έτσι εξασφαλίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίασή του και προσβλέπω στην εξέτασή του φακέλου κύκλο τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you. Now for Aldi, Sophie. Ευχαριστώ και τώρα για τον Άλντι Σόφη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζω την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει Απλώς ήθελα να κάνω κάποιες ε, επιμέρους παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το γενικότερο θέμα του ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θα πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτό το είδο τα ζητήματα, εγώ πιστεύω πως ναι. Δεν θα καθορίσει τα συστήματα που τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν μεν, αλλά από καιρό, από πολύ καιρό, με το Σύμφωνο Σταθερότητα έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι έχουμε την υποχρέωση να είναι βιώσιμα τα συνταξιδοτικά μα συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει κάθε δικαίωμα να εκφραστεί όχι μόνο για τι λεπτομέρειε των συστημάτων, αλλά κυρίω για την βιωσιμότητά του. Για τι κεφαλαιοχικέ απαιτήσει, για πολλά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου, εκφράστηκαν ανησυχίε. Ανησυχίε εκφράστηκαν βέβαια και από τον εισηγητή, και από τον ε, Σκύο συγκεκριτή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σε μεγάλο βαθμό είναι δικαιολογημένες, αλλά εδώ υπάρχει και ένα χάσμα το οποίο το παραβλέπουμε. Αυτή η αντίσταση στο θέμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν είναι λίγο κοντόφθαλμη. Διότι αν αποδεχτούμε τον κίνδυνο αν αποδεχόμαστε μάλλον τον κίνδυνο, ίσως τελικά ο κίνδυνος αυτός ε, να εξαπλωθεί σε βαθμό καθόλου ισότιμο μεταξύ των διαφορετικών γενεών, των διαφορετικών ηλικικών ομάδων. Μήπως τελικά το βάρος το αναλάβουν οι μελλοντικές γενιές. Αυτή είναι μια υποχρέωση που πρέπει να την... Αυτή... Είμαστε υποχρεωμένοι να το σκεφτούμε αυτό. Ή μιλάμε για την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη προς τους συνταξιούχους, όμως αλληλεγγύη πρέπει να είμαστε και προς τις νέες γενιές, που θα γίνουν κάποτε συνταξιούχοι του μέλλοντος. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε λίγο πιο ανοιχτό πνεύμα στην έκθεση. Το είπατε κι εσείς νομίζω, προς τις ε, επιμέρους της ε, λύσεις που θα είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένα θέματα. ας δούμε και τι γίνεται με τους εργασιακούς κύκλους. Δεν διαβουλεύουν πια οι άνθρωποι 40 χρόνια για τον ιδιοκοδότη σε μεγάλες βιομηχανίες πλέον. Έχουμε ένα εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι μέλη εργατικού συνδικάτου. Και πολλές επιχειρήσεις ε, είναι ιδιοκτήτες συνταξιδοτικών ταμείων, δηλαδή οι ίδιοι συνεισφέροντες είναι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πως έχουν διαμορφωθεί σύγχρονοι εργασιακοί κύκλοι. Και για το διασυνοριακό ζήτημα. Λέτε ότι μόνο το 3% το 3% των πολιτών μπορεί να μεταθέλουν να μεταφερθούν ως συνταξιούχοι σε άλλο μέλος. Όμως, είναι πολύ περίεργο να μην μπορεί κανείς να μεταφερθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασκήσει το επάγγελμα που θέλει, να εξασκήσει την ελεύθερη κινητικότητα. Εδώ στέλνουμε ανθρώπου στη Σελήνη ή όπου θέλουμε. Είναι πολύ κακό να είναι αποτρεπτική η θεμελίωση συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν τα κάτι μέλη θα πρέπει να κάνουν κάτι και να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που κρεμεί εδώ και τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. Um, for the Greens. Από τους Πρασίνους ο Φιλί Λαμπέρτς. Καλημέρα σας και πάλι. Μερικά σχόλια. Καταρχάς συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι σημαίνει πρώτος, δεύτερος και τρίτος πυλώνας, γιατί σε διαφορετικές χώρες σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν ορισμό για να συγκρίνουμε όμοια μεταξύ τους πράγματα. Και επίσης οι ποιοτικέ προδιαγραφές για την εταιρική διακυβέρνηση, τη δίκηση επιχειρήσεων και όλα αυτά ε, είναι σημαντικά. Είναι ένα τομέα που θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πιστεύουμε και το λέω γιατί αυτό το καιρό εργάζομαι και για τους ε, Ευρωπαίους πράσινους για αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε, λέω, μια σοβαρή ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τα συνταξιδοτικά συστήματα στα 27 κράτη-μέλη, μια σοβαρή μελέτη, να μάθουμε τα στοιχεία. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά έγγραφα σχετικά, αλλά εγώ ακόμα δεν έχω δει ε, συγκριτική μελέτη σε βάθος των συνταξιωτικών συστημάτων στην Ένωση. Που είναι το πρώτο βήμα θέλουμε να κάνουμε κάτι από κοινού ή να φρονούμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Εκεί που διαφωνούμε με τον εισηγητή είναι η απόρριψη της κοινοτική νομοθεσίας για τα ποσοτικά στοιχεία ε, των ε, συνταξιωτικών ρυθμίσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια ενιαία αγορά. Δεν είναι μόνο ένα έμβριο πολυεθνικής δημοκρατίας, αλλά είναι και ένας χώρος κοινών, κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτή τη στιγμή δεν αρκούν αυτά. Και επίσης αυτό εξηγεί και τις διαιρέσεις που βλέπουμε στην Ευρώπη αυτό τον καιρό. Προφανώς δεν θέλουμε σε ένα ενιαίο σύστημα ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης. Δεν ξέρω αν το επιθυμεί και κανείς αυτό. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε κοινά βασικά δικαιώματα. Ε, είναι τα θεμέλια, αν θέλετε, ή μια πρώτη στιβάδα της κοινή κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό έχει σημασία. Γιατί αν θέλουμε να δημιουργήσουμε όχι μόνο την αίσθηση, αλλά την πραγματική έννοια ότι δεν έχουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Ευρώπη, έχουμε όλοι τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα. Και δεύτερο, ε, αν θέλουμε να απορροφηθούν οι κραδασμοί, ε, ε, που υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το σύστημα απορρόφηση κραδασμών, γιατί ο κόσμο δεν μπορεί να κυκλοφορεί τόσο ελεύθερο και να εργάζεται, ε, γιατί δεν μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά του από τη μια χώρα στην άλλη. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ, ελάχιστα συνταξιωτικά δικαιώματα. δεν μπορεί να είναι σε θέση η Ευρώπη να το κάνει αυτό. Επίση, διαφωνούμε με τον εισηγητή στο θέμα της εναρμόνισης ε, των προδιαγραφών προληπτικής εποπτείας και αν αυτό είναι βλαβερό. Ειλικρινά έχω ενοχληθεί, για να μην πω ότι έχω εξοργιστεί από κάποιους που λέγουν ότι θα κάνουμε διάφορα πράγματα για τις τράπεζες, αυτό θα αυξήσει το κόστος δανειοδότησης. Κάνουμε πράγματα στη συντάξη, αυτό θα αυξήσει το κόστος των εισφορών. Έχω βαρεθεί να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ε, ε, είναι, ε, φαίνεται λιγότερο δαπανηρό βραχυπρόθεσμα όταν κάνουμε τσαπατσουλιές και γρήγορα γρήγορα προσπαθούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Αν θέλουμε να τα λύσουμε με τρόπο συστηματικό και κανονικό και τα συνταξιδοτικά, είναι λάθος αυτό που προτείνεται και θα πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα και ο κίνδυνος έχει το τίμημά του. Και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο θα πρέπει να ε, βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Έχω βαρεθεί αυτή την οτροπία. Δεν υπάρχουν τζάμπα γεύματα. Το τζάμπα έχει πεθάνει. Λοιπόν, τα πάντα έχουν το κόστος τους και θα πρέπει να το αναλαμβάνουμε. Τώρα, ε, το τι ε, σημαίνει ε, σύνταξη επαρκής ασφαλής και βιώσιμη, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσω. Και βέβαια δεν έχω καμία αντίρρηση να έχουμε δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης ιδιωτικά ε, κεφαλαιοποίησης, ε, ανταποδοτικά. Ε, όπως και στις τράπεζες και στις συντάξεις και στα συστήματα χρειάζεται ποικιλία για να είναι και πιο ανθεκτικά τα συστήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που εμείς ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι η βασική κύρια σύνταξη που να αντέχει στη φτώχεια. Ε, δεν μ' να μιλάω για πρώτο πυλώνα γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είναι σύγχυση με τους πυλώνες. Ε, το κράτος θα πρέπει να εγγυάται αυτό το δικαίωμα τη βασική σύνταξη κατά τη φτώχεια, το ελάχιστο εισόδημα. Τώρα, αν κάποιο άλλο θέλει να έχει μια επικουρική σύνταξη ε, ιδιωτικά ή με την επιχείρησή του, καλώ. Και έρχομαι τώρα και απευθύνομαι σε εκείνου που ζητούν η εξηγένση των δημοσίων οικονομικών. Αν θα πρέπει τα δημόσια χρήματα να πηγαίνουν στην υποσύρριξη των συντάξεων, αυτό θα πρέπει να είναι η βασική κύρια ε, ε, σύνταξη και δεν δέχομαι να επιδοτούμε με πενιχρούς πόρους βασικά ιδιωτικά συνταξιωτικά συστήματα που είναι άνισα και από το σχεδιασμό τους Καλά, εντάξει, πάντα υπάρχει ένα επίπεδο ανισότητας, αλλά εκνά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει δημόσια κονδύλια βασικά να ε, επιδοτούν τους πιο εύπορους στην κοινωνία. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο και ε, ε, συμβαίνει ευρύτατα, περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτοί που ζητάτε περικοπές στι δημόσιες δαπάνες, για να δούμε τι έχετε να μα πείτε. ακριβώ οι ίδιοι θα βγείτε στα οδοφράγματα ε, για ε, να υπερασπιστείτε αυτές τις καταστάσεις που ευνοούν ευπόρους. Ε, καλή την πίστη. εντάξει, μπορεί κάποιος να ζητάει περικοπές. Αλλά θα ήθελα να δω την ίδια αγωνία για περικοπές και σε αυτούς τους τομείς, γιατί όσοι ζητάνε ε, να κοπούν επιδόματα ανεργίας και άλλα κοινωνικά επιδόματα. Τότε ε, θα πιστέψω στην καλή του πίστη. Μέχρι να το δω όμως αυτό, ε, θεωρώ ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ευχαριστώ. Ο Σαΐντ. Σαϊντ, συγγνώμη. Um, how do I follow Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα προσπαθήσω να μιλήσω σε διαφορετικό πνεύμα και να σας κάνω λίγο πιο ευχάριστο το κλίμα. Καλωσορίζω τις προτάσεις του εισηγητή. Δεν έχω πολλά να επισημάνω προς το περιεχόμενο. Είναι σαφές ότι ο πρώτο και ο δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως θα πρέπει και εμείς να παρακολουθούμε τι γίνεται και να έχουμε πολύ ανοιχτό πνεύμα. Να ακούμε όσους λένε ότι θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρονται τα συνταξιδοτικά δικαιώματα χρειάζονται συνένεση ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινή αγορά και να διευκολύνουμε την κινητικότητα των εργαζομένων, των πολιτών. Όμω ταυτόχρονα θέλουμε να διατηρήσουμε και την αρμοδιότητα στα κρατημέλη. Πώ θα μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά των συντάξεων δικαιωμάτων. Επίση, συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι πρέπει να έχουμε υπόψη και την νομική βάση. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα και όχι να υπάρχει ένα θέμα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων και διακλειστίδας αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σα πω τώρα, εγώ με τι έχω κουραστεί, όπως είπε και ο προλαλή σα. Έχω κουραστεί να διασώζουμε τις τράπεζες στο ΕΒ Βασίλειο μετά τη Lehman Brothers και να έχουμε τόσα νομοθετικά μέτρα, αλλά να μην έχουμε επιλύσει το δεμελιώδε ζήτημα του συνταξιδοτικού μας συστήματος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα χρειαστεί πάλι οι φορολογούμενοι να απομιστούν τις ευθύνε και το τίμημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περάσει και εκείνη αυτό το θέμα σαν μια κρίση όπου θα πρέπει να έχουμε καλύτερες ρυθμίσεις για περισσότερη Ευρώπη. Και επειδή εδώ μιλάμε για συντάξεις, να πω ότι ανησυχώ για την υλοποίηση του Φεραγγιώτα 2 του Σόλβενση δύο όπως και ο εισηγητής, και νομίζω ότι πρέπει να ακούμε όσους λένε ότι θα ξεφύγουν, θα, θα διατρέξουν τα χρήματα για τις τράπεζες. Και εγώ συμφωνώ, ούτε εγώ τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Διότι αν δεν είχαμε τους ισολογισμούς τους να προσέχουμε δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα τώρα. Εάν ίσχυε η προληπτική υποπτία θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα υπήρχαν τέτοιε απώλειε και δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να δίνουμε ευήκονους όταν θέλουμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των συνταξιδοτικών συστημάτων και των εταιριών ασφαλίσεων ζωής. Μπορεί δισεκατομμύρια ευρώ να ξεφύγουν από την πραγματική οικονομία και να φτάσουν στα χέρια αυτών των εταιριών ουσιαστικά. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Συνένεση. Είδαμε να υπάρχει όχι μόνο από του εργοδότε, αλλά και από, τα, από τι συνδικαλιστικέ οργανώσει των εργαζομένων που ανησυχούν για τα συνταξιδοτικά συστήματα και τι συντάξει του. Θέλουμε να αναλάβουν οι πολίτε την ευθύνη για τη δική του ε, σύνταξη. Όμω, θα πρέπει και εμείς κάτι να τους εξούμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Κάποιοι που κερδίζουν μικρά ποσά ουσιαστικά βρίσκονται σε δυσχερή θέση γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις εισφορές για τη σύνταξή τους. Εκεί το κράτος μπορεί να παράσχει αυτή την υπηρεσία. Απλώς ας παροτρύνουμε όσο μπορούμε τους πολίτες να αναλάβουν ευθύνες για το δικό τους μέλλον. Κάποιοι ούτω ή άλλω έχουν ξεχάσει ότι θα μπορούσαν να έχουν την ίδια δουλειά για μια ζωή. Δεν μπορεί να δουλεύουν για, για την ίδια εταιρεία, για τον ίδιο οργανισμό. Κάποιο που δουλεύει στου σιδηροδρόμου, ε, στο, στα λεωφορεία, ξέρει ότι μπορεί να μην ολοκληρώσει τον εργασία του κύκλο. Εγώ έχω αλλάξει αρκετέ θέσει εργασία και άλλαζα τη σταδιοδρομία μου και την κατεύθυνσή τη ανάλογα με τι ευκαιρίε. Οι άνθρωποι τώρα το κάνουν αυτό όλο και περισσότερο. Με την αλλαγή σταδιοδρομία, με τη διαβίου μάθηση. Θα πρέπει λοιπόν με την αλλαγή στον τόπο που εντοπίζουν τη δραστηριότητά του, θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν και τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα. Ακούσαμε με την προληπτική εποπτεία τη Γερμανία ε, και πόσο καλό ήταν αυτό το παράδειγμα. Θα πρέπει και εμείς να διδαχθούμε από αυτό. Για να συνοψίσω λοιπόν, νομίζω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Και όπου παρέμβει, να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ζημιώσει τα εθνικά συνταξιωτικά συστήματα. τα οποία ε, πολλές φορές είναι βαθιά ριζωμένα στην πολιτική και οικονομική και κοινωνική νοοτροπία που επικρατεί στις χώρες τους. Πάντως ευχαριστούμε τον εισηγητή και θα είμαστε στη διάθεσή του για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος παρακαλώ. Ο Πίτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Είμαι, ήμουν εισηγητής για την αφαιρεγγιότητα 2 πριν από πολύ καιρό και ξέρετε ότι όλα κρίνονται από αυτά που θα πούν οι άνθρωποι, άσχετα με το αν έχουν γίνει οι σωστοί υπολογισμοί. Χρησιμοποιούν κάποιοι ε, την φρεγιότητα 2 για την, τον σχεδιασμό των συνταξιδοτικών συστημάτων ε, ή όχι. Κάποιοι το είχαν προβλέψει, κάποιοι άλλοι όχι. Και το συνδυάσαν και με τις κεφαλαιακές απαιτήσει. Υπάρχει και η οδηγία για τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής δέσμη, IOP. Οπότε Υπάρχουν 1.400 διαφορετικά προϊόντα για ασφάλεια ζωής και είναι δεκαπλάσιος ο αριθμός για τις ασφαλιστικές συντάξεις. Εννοείται ότι συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Πολλές ε, οι ισχύουσε συνταξιδοτικέ ρυθμίσει ε, καλύπτονται από τον κοινωνικό διάλογο. Είτε μα αρέσει είτε όχι, όμω υπάρχουν και τα μαύρα βιβλιαράκια και προηγούμενε ρυθμίσει που ό,τι και να αποφασίσουμε εκείνοι θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο. Και μπορεί να αληθεύουν αυτά που μα λέει η Σοφή. Υπάρχει και το SCR στην φαρεγγιότητα 2, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να είναι κάποιος επικριτικός, αυτό δεν με ενοχλεί, αλλά πραγματικά αν λέτε ότι όχι θα μαυρώσουμε την εικόνα της φερεγγιότητας 2 και ότι αποκλείεται να λειτουργήσει το σύστημα, δεν θα προχωρήσουμε. Ας δούμε στις αξιωτικές ρυθμίσεις μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, όπως πρέπει να γίνει και για τα ε, επενδυτικά προϊόντα λιανικής. Ε, θα χρειαστεί σε πρόωρο στάδιο συνεργασία όλων, αλλά ξέρετε, είναι ένας αγώνας χρόνου. Πρόκειται για μακροπρόθεσμα προϊόντα, αλλά χρειαζόμαστε τη σωστή βάση. Ε, ας είμαστε όμως ξεκαθαροί, σε κάθε τομέα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προσδοκίες για τα αναμενόμενα αποτελέσματα, για τις εισφορές, για τις παροχές των διαφόρων ασφαλιστικών συστημάτων και πραγματικά υπάρχει ένα ε, στοιχείο ε, κρατικού φορέα, δηλαδή θα πρέπει όταν οριμάσουν κάποια από αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα να καλύφθει ένα κομμάτι από τα κράτη, αλλά όχι μόνο. Ε, εδώ πιέζουμε τους ανθρώπους να ε, υπογράψουν ιδιωτικές ασφάλειες. 60% του, του εργατικού δυναμικού στην Ιρλανδία, κάποια στιγμή θυμάμαι, ε, μετά από παρότρινση της κυβέρνησης είχε υπογράψει τέτοια, τέτοιες συμβάσεις τρίτου πυλώνα, ατομικής σύνταξης. Και τι θα γίνει, κάποια στιγμή θα τους ανακοινώσουμε ότι όχι, θα πάρετε λιγότερα λεφτά, παρότι εσείς είχατε υπολογίσει και είχατε συνεισφέρει για παραπάνω. Δεν γίνονται αυτά επίσης με τη γύρανση του πληθυσμού. Ε, πρέπει να καταλάβουμε τι θα κάνουμε με το όριο της φτώχειας. Θα πρέπει να προβλέψουμε τώρα τι θα κάνουμε με τα προβλήματα και όχι να τα αφήσουμε για μετά. Επίση, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την προσέγγιση που τελικά θα υιοθετήσουμε. Καλωσορίζω εν γέννη λοιπόν την έκθεση του Τόμας. Ε, ακόμη πολύ σοβαρό έργο. Ας ακολουθήσουμε ε, τις συμβουλές κάποιων ρυθμιστικών οργάνων σε σχέση με την προσέγγιση τους ε, μέχρι στιγμής, αλλά να γνωρίζουμε ότι θα γίνει σκληρό αγώνα ανάμεσα στα ίδια τα κράτη-μέλη που θέλουν να εξασφαλίσουν ε, την ε, ποιοτική αντιστοιχία ανάμεσα στα συνταξιωτικά και τα ασφαλιστικά συστήματα. Μα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι που ε, είναι προετοιμασμένοι να χρησιμοποιήσουν τα ασφάλεια ζωής για να μπορέσουν να πληρώσουν τις συντάξεις στου εργαζόμενου του. Οπότε τώρα ίσω κληθούν να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει φερεγγιότητα 2. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το υποστεί ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και να ειδοποιήσουμε ότι η φερεγγιότητα 2 δεν θα ενταχθεί στην IORP και δεύτερον τα μεμονωμένα κράτη-μέλη δεν τα να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς περιμένουν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη να κάνει το ίδιο σφάλμα με εκείνους. Δεν χρειάζεται. Σα ευχαριστώ, άλλος κανείς. Μερικά σχόλια από πλευρά μου. Ευχαριστώ πρώτα απ' που αναγνωρίζετε ε, αυτό το έργο και αυτό τον αγώνα που κάνουμε με άλλες επιτροπές για τις αποκλειστικές ε, αρμοδιότητες ε, δεν είναι ότι δεν έχουμε δουλειά και ψάχνουμε αλλά όταν μπαίνει στα χωράφια μας μια άλλη επιτροπή θα πρέπει να επέμβουμε και το κάνουμε κάθε φορά και ευχαριστώ και τη γραμματεία τον τους δύο παρακαθήμενους εδώ, ε, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο αυτή η υπόθεση, η οργάνωσή της και ο ε, εντοπισμός του που βρίσκονται οι δικές μας αρμοδιότητες. Συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο Πίτερ, αλλά αυτό δεν θα σας εκπληξεί, γιατί ήμουν σκιώδης εισηγήτρια στη δική του έκθεση για τη 2. Όταν ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά των συνταξιούχων, πρέπει να ξέρουμε ότι και τα συνταξιωτικά ταμεία ε, είναι μεγάλοι επενδυτές στην οικονομία και όταν αρχίζουμε και ανακατεύουμε τις κεφαλαϊκές τους απαιτήσει, επηρεάζει αυτό όχι μόνο τις συντάξεις αλλά και την οικονομία την ίδια. Το είδαμε αυτό και στη Φερεγκιότητα 2 ε, χρειάστηκε με την με Omnibus 2 να ε, επικυρωποιηθούν όλα αυτά. Βέβαια στην Ευρώπη έχουμε κρίση οικονομικής μεγέθυνσης και τώρα η ε, ρυθμιστική ανασφάλεια επιτείνει την κρίση σε μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει τώρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να πούμε τερματίζουμε αυτή την ανησυχία και την ανασφάλεια γύρω και μέσα στα συνταξιωτικά ταμεία στην Ευρώπη, τα ιδιωτικά. Ε, και ε, καλά κάνουμε και έχουμε αυτή την έκθεση γιατί αυτό βοηθάει την οικονομία. Ε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο ως κοινοβούλιο και νομοθέτης να πούμε ότι όλα θέλουμε απολύτως να είναι κλειδωμένα και θωρακισμένα, να μην έχουμε καθόλου αγορές για να μην υπάρξει επόμενη κρίση γιατί βρισκόμαστε επικίνδυνα ε, κοντά σε όλα αυτά, πολύ επικίνδυνα με όλες αυτές τις διαδράσεις και την επιρροή της μιας νομοθεσίας ε, στην άλλη. Βεβαίως και θέλουμε να προστατεύσουμε τις συντάξεις και να μην χάσει κανείς τη σύνταξή του, αλλά ο καλύτερος τρόπος να είναι να είναι τέτοια η απόδοση που να μην έχουν ποτέ ε, αξιοπρεπή σύνταξη και να είναι τόσο χαμηλά τα επιτόκια στα ομόλογα ώστε ο κόσμος να αγωνίζεται για να αποκομίσει ένα εισόδημα. Λοιπόν, ε, κάποια στιγμή ε, να πούμε stop μέχρι εδώ, να μην επιδεινωθεί άλλο η κατάσταση. Για τα γενικά σχόλια σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά ευχαριστώ Τόμας και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε αυτό σας δίνω και πάλι το λόγο. Äh, Ευχαριστώ πολύ Σάρον και τους συναδέλφους για τα σχόλια, για τη συμφωνία αλλά και τις ε, κριτικές ε, παρατηρήσεις. Το πλεονέκτημα ε, στο Κοινοβούλιο είναι ότι γνωριζόμαστε και πάνω κάτω και μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα πάει η συνεργασία. Είναι δεδομένες οι προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, στα κράτη-μέλη έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Έχω κάνει συζητήσεις εδώ στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν κατάλαβαν κάτι που ισχύει στη Γερμανία. Είπαμε να έχουμε συστήματα εταιρικών συντάξεων που ισχύουν και είναι ε, βιώσιμα. Δηλαδή, ε, θέλουμε να επιβραβεύσουμε κάποιον που είναι ε, πιστός στην εταιρεία. Υπάρχουν χώρες που αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Δεν θέλουμε... <laughs> Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν, ούτε να μην τον αφήσουμε να έχει κινητικότητα, αλλά θέλουμε να επιβραβεύσουμε κάποιον που παραμένει στην εταιρεία ε, και ε, φροντίζει ε, να ενισχύσει και με το Ταμείο το Συνταξιδοτικό. Κανείς δεν πρόκειται να μείνει ή να φύγει από μια εταιρεία λόγω αυτού του επικορικού ταμείου του εταιρικού. Και τα συνταξιωτικά δικαιώματα δεν χάνονται, συνυπολογίζονται. Η πίστη λοιπόν στην εταιρεία είναι σημαντικό για μας και δεν είναι καθόλου εμπόδιο στην κινητικότητα. Δυστυχώς ορισμένοι κύκλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι το ερμηνεύουν και λυπούμε εγώ γι' αυτό πάντα. Δεν ξέρω μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε. Και βεβαίω είναι σημαντική η βιωσιμότητα. Κοίταξτε στη Γερμανία, οι εταιρικέ συντάξεις είναι 460 δισεκατομμύρια ευρώ, τεράστιος μηχανισμός διάσωση. Εκεί να δείτε πόσε χώρες μπορούμε να διασώσουμε. Γιατί είναι ε, σημαντικό να διατηρηθεί αυτό. Γιατί τώρα είναι μηδενικά τα επιτόκια στην Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή. Για ρωτήστε εκείνους που διαχειρίζονται αυτά τα συστήματα ε, πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθούν. δεν μπορούμε να θέλουμε τέτοια κατάσταση. Στην Ολλανδία έχετε θαυμάσιο σύστημα και ένα τεράστιο τομέα, ε, πολλαπλάσιο του γερμανικού και το γνωρίζω και από την εισηγήτρια. Ε, θα πάω στην Επιτροπή Απασχόλησης τώρα που ε, ε, το συζητάει και θα συζητήσουμε και με την ε, εισηγήτρια της έκθεσης ε, πρωτοβουλίας. Έχει σημασία και ελεγγύη με τις νέες γενναίες. Αλλά όταν κάποιος μπαίνει στην αγορά εργασίας θα πούμε ότι θα πρέπει να μείνεις λίγο καιρό στην εταιρεία για να έχεις δικαίωμα σε σύνταξη. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε ένα job hopping, να, να, φεύγει από τη μια εταιρεία να τρέχει στην άλλη και να χρηματοδοτείται και συνταξιδοτικά. Θα πρέπει να αξίζει τον κόπο αυτό το σύστημα. Δηλαδή έρχονται οι νέοι, μπαίνουν λίγο καιρό, μένουν λίγο καιρό στην εταιρεία και ε, δεν μπορεί να σταθεί το σύστημα όταν σηκώνονται και φεύγουν. Δεν θέλουμε, εμεί θέλουμε βιώσιμο, βιώσιμο σύστημα. Ο συνάδελφο Ναμπέρ των Πρασίνων έχει ήδη αποχωρήσει και βέβαια έχει δίκιο, έχει την τιμή του και ο κίνδυνο. Αλλά σωστό είναι, αλλά σε ποιο βαθμό θα πρέπει να υπομισθούμε εμεί. Δεν θέλουμε κοινωνία δύο κατηγοριών. Ποιο το θέλει εδώ μέσα, κανεί. Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε συστήματα που να μπορούν να χρηματοδοτούνται σωστά, αλλά να πούμε να μην τα κάνει όλα η Ευρώπη. Ένα συνάδελφό μα έχει αλλάξει 5-6 δουλειέ και μετά έγινε βουλευτή. Ελπίζω στο μέλλον να μην σου κόψουμε την καριέρα και να μπορέσει να έχει άλλε 5-6 θέσει. Κανεί δεν είναι μονοδιάστατος. θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους νέους και τους πιο ε, μεγάλους σε ηλικία να ε, ε, βρίσκονται σε ένα σύστημα με λογική και σωστή χρηματοδότηση και να έχει νόημα αυτό το σύστημα και το, της εταιρικής σύνταξης. Εσύ, Πίτερ, είχες μακρά εμπειρία και είχαμε και καιρό να το πούμε στη η Βρετανία ξέρουμε ποιο είναι το σύστημα και είναι καλή χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να συγκριθεί η ασφάλεια ζωής με τα συνταξιδοτικά συστήματα. Είναι τελείως διαφορετικό. Το stress test τελείωσε και το περάσαμε επιτυχώς. Ε, γιατί έχουμε καλές δομές ε, βιώσιμες και λειτουργικές. Τέλος, ευχαριστώ και τη Σάρων και τη Γραμματεία, γιατί πραγματικά ε, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι, πέρα από τις ίδιες αρμοδιότητες που έχουμε εμείς στην Οικονομική Επιτροπή, είναι και καλή συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης. Λοιπόν, φεύγω και πάω εκεί και με αυτή τα καλά νέα ε, και χαίρομαι ε, για τη συζήτηση που θα κάνουμε με τους Κιώδης και τα άλλα μέλη. Είναι μια πολύ καλή αφετηρία και βάση ε, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλό ισόρροπο αποτέλεσμα. Βέβαια για μια ελπίδα ζούμε και όλοι ξέρουμε ότι είμαστε δυναμικοί συνάδελφοι και εργατικοί και νομίζω ότι θα φέρουμε αυτή την υπόθεση σε αίσιο πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Δυστυχώς είναι πολύ στενές προθεσμίες εδώ. Για την υποβολή τροπολογιών 11 Δεκεμβρίου, εξέταση του σχεδίου έκθεσης 10 Ιανουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Ιανουαρίου και στην Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή 23 Μαρτίου, ενώ στην 21 Μαρτίου, ενώ στην Ολομέλεια θα περάσει τον Απρίλιο για την εξέταση των τροπολογιών. Καλό θα ήταν να υποβληθούν τροπολογίες μόνο σε ό,τι αφορά το τμήμα όπου έχει είτε αποκλειστική είτε μεικτή αρμοδιότητα η Επιτροπή μας. Εάν θέλετε να πείτε κάτι για τα άλλα υπόλοιπα τμήματα της έκθεσης, ξεχωριστές τροπολογίες παρακαλώ. Μην μπερδευτούν με εκείνα όπου έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα ή καμία αρμοδιότητα. Διότι τότε Μπορεί να τα δει όλα η Επιτροπή Ασχόλησης και να μην διατηρήσουμε την δική μας αποκλειστική αρμοδιότητα. Αυτό να το έχουμε κατά νου γιατί και η γραμματεία και ο Συγκριτής θα πρέπει να ασχοληθούν και να ετοιμάσουν συμβαστικέ τροπολογίες. Να είναι σαφεί λοιπόν οι κατηγορίες αποκλειστική αρμοδιότητα τη Επιτροπή Οικονομικών και Νοσματικών Υποθέσεων και εκεί να ψηφίσουν ξεχωριστά. Τα υπόλοιπα να είναι λίγο παράμερα. Θα είναι χρήσιμο νομίζω και πιστεύω αυτό θα ήταν ο καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε και να συντάξετε τι τροπολογίε σα. Ευχαριστώ λοιπόν. Νομίζω δεν υπάρχουν διάφορα και ο συνήθω θα συναντηθούμε στο Στρασβούργο στι 10 Δεκεμβρίου. Δεν νομίζω να κρατήσει πολύ πάντως εκεί η συνάντηση. Ναι. Ζαν Πολ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να μην σα καθυστερήσω επειδή είναι και αθρώα η προσέλευση. Απλώς ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στις 11 στην διάσκεψη των πρόεδρων θα μιλήσει για τη δημιουργία μιας ειδική επιτροπής για την Ευρωζώνη. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί της ουσίας, αλλά από την σκοπιά της μεθόδου είναι περίεργο να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα στην ε, Επιτροπή μας παροσκηνιακά. Ε, μοιράστηκε το σημείο με αυτό του Προέδρου σε ορισμένα μόνο πρόσωπα και θα έπρεπε το Κοινοβούλιο να μπορούσε να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Και έχει τοποθετηθεί γιατί επί της έκθεση της κυρίας Μπερές για την κρίση είχε γίνει αυτή η πρόταση στα πλαίσια της δικής μας της Επιτροπής να δημιουργηθεί μια υποεπιτροπή για να διαχειριστεί τα θέματα της κρίσης, πρόταση η οποία δεν προκρίθηκε. Επιπλέον πρόσφατα με την αφορμή της έκθεσης Tyson το θέμα τέθηκε ξανά και φάνηκε ότι στο κοινοβούλιο αυτό η πλειοψηφία τέλο πάντων των βουλευτών που ασχολήθηκαν με την έκθεση αυτή ήταν κατά μια τέτοια εξέλιξη που δεν θα επέτρεπε στο κοινοβούλιο να αναλάβει σωστά τι αρμοδιότητέ του και δεν θα είχε και νομική βάση. Τελικά επανέρχεται όμω το θέμα. Βάσει των όσων γνωρίζω, δεν έχει εκτελεστικέ αρμοδιότητε όμω ο πρόεδρο του κοινοβουλίου. Και Όσοι μιλούν για δημοκρατικό έλεγχο διαρκώ, καλά θα ήταν να τον εφαρμόζουν κιόλα όταν πρόκειται για το ίδιο το θεσμικό μα όργανο. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, θα σα παρακαλέσω το θέμα αυτό να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών τη Δευτέρα το βράδυ. Διότι καλό θα ήταν να το μελετήσουμε το θέμα. Λυπάμαι, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς ενημερωθήκατε, ε, όπως και πολλοί από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και αυτό δείχνει μια περιφρόνηση προς τα πρόσωπά μα συμπεριλαμβανομένης της Προεδρίας προς τους βουλευτές. Στιγμές δύσκολες για την Ευρώπη, στιγμές όπου δεν θα έπρεπε, θα είναι ανόητο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κάποιες υπηρεσίες, ε, υπηρεσίες που κάνουν προτάσεις τις οποίες δεν θέλησε το ίδιο το Κοινοβούλιο. Για την εκπροσώπηση τη Ευρωζώνης σίγουρα υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και πιέσει του Συμβουλίου ώστε να μην υπάρχει συμμετοχή του, Ευρωκοινο... του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά αν διαβάσει κανεί το σημείωμα είναι πολύ άκομψο. Οι Βρετανοί φίλοι θα εκπλαγούν που το ονομάζω έτσι. Ε, με τρόπο άκομψο απομακρύνονται και οι Βρετανοί φίλοι από, τους, ε, από την όλη συζήτηση. Ξέρετε ότι δεν είμαι παθιασμένο στο θέμα αυτό δεν είμαι αγγλωμανή, αλλά σε ένα κλαμπ που όλοι είναι μέλη θα πρέπει να είναι ισότιμη και ώρα του παιχνιδιού. Ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Και εγώ δεν το έμαθα απευθεία, αλλά το άκουσα από, από το Σφέν και του είπα αμέσω ότι θα το προβλέψω στην συνάντηση των συντονιστών της Δευτέρας. Εν όμως και εγώ σημειώνω, στέλνω σημειώματα και ενημερώνω γιατί αυτό αντίκειται με όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής μας. Επιβεβαιώνω ότι η δική μας γραμματεία της Επιτροπής ΕΚΟΝ δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό. Είναι πολύ ανητικό να μην γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτά και κανείς δεν έμαθε τι συνέβαινε. Είναι πολύ σοβαρό και όπως είπες Τώρα να λέμε να γίνει μια επιτροπή που επιτροπή να συμμετέχουν όλοι όσοι είναι στο ευρώ ή μπορεί να μπουν στο ευρώ και πρόσωποι της Δανίας, τέτοια επιτροπή αντίκειται στις αρχές της της συνθήκης. Δεν μπορεί να έχει νομοθετικές ε, αρμοδιότητες. Ίσως κάποτε στο απότερο μέλλον, όταν θα υπάρχει περισσότερος δημοσιονομικός συντονισμός, όταν αλλάξει η συνθήκη, ίσως κάτι τέτοιο να ανακύψει ως ανάγκη, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Επίσης, το σημείωμα νομίζω παρανοεί τελείω την ε, σχέση μεταξύ του τι ισχύει για την εποπτεία και το τι πρέπει να γίνει στην ενιαία αγορά, τις κεφαλαιακές απαιτήσει, τα δευτερογενή μέτρα που θα που θα προέλθουν από την, ε, για την τραπεζική αρχή με το κοινό ε, εγχειρίδιο και τους, ε, τις αλλαγές στον κανονισμό EBA για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Όλα αυτά είναι στο επίπεδο της, ενισα... της ενιαίας αγοράς. Θέλουμε εναρμόνιση και όχι κάτι διαφορετικό. Το βρίσκω λοιπόν πολύ παράξενο Ενώ είναι σαν να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει opt-out στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν ποτέ να έχουμε αυτές σε αυτό το σημείο. Πίτερ, ε, τη Δευτέρα στο Στρασβούργο ε, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Οι συντονιστές έπρεπε να το συζητήσουν αυτό το θέμα ε, κανονικά, αλλά αν θέλουμε ευρύτερη συζήτηση πρέπει να είμαστε όλοι. Σάρον, συμφωνώ. Αλλά όπως ήδη είπα από πλευράς Επιτροπής, έχουμε αποφανθεί από αυτού τουλάχιστον τρεις φορές ε, μετά από συζήτηση, αλλά θα το χώσουμε και αυτό στην ημερήσια διάταξη, αν χωράει, για να ενημερωθεί και η Επιτροπή για τα όσα διαμείβονται στη διάσκεψη των Προέδρων. Ζαν Πολ, σε ευχαριστούμε που έθεσε το ζήτημα και ε, θα το παρακολουθούμε. Τα λέμε στο Στρασβούργο.